Καλημέρα συνάδελφοι. Ευχαριστώ που ήρθατε στην ε, δεύτερη φετινή συνεδρίαση. Έχουμε διερμηνία που τη ζητήσατε και θα έχουμε και βίντεο διάσκεψη με τις Βρυξέλλες. Any objections to the draft agenda? Έχετε αντίρρηση στον φάτο το σχέδιο μερίσιας διάταξης. Δεν βλέπω. Εγκρίνεται. Αντιρρήσεις στον αφορά το σχέδιο πρακτικών. Εγκρίνονται ανακοινώσεις δεν φαίνεται να φέραμε τύχη στον Gordon Sandland που ήταν τόσο καλός ε, ομιλητής στην προηγούμενη σύνοδο. Έχασε την εμπιστοσύνη του Προέδρου του και ανεκλήθη από τη θέση του. Ο Μαρκ Λίμπη, ο επιτετραμένος της Αμερικανικής Αποστολής, ήταν ομόλογός μας, μέχρι να αλλάξουν τα πράγματα και θα περιμένουμε μέχρι τουλάχιστον τέλος του έτους με να γίνουν εκλογές, η, διαδικασία της γερουσίας. Δεν θα περιμένουμε καινούριο πρέσβη πολύ σύντομα. Μετά την αναχώρηση της κυρίας Τζάκι Τζόουνς πρέπει να διορίσουμε μια γυναίκα σαν δεύτερη αντιπρόεδρο και θα το κάνουμε αυτό στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Τη συνεδρίαση της 6ης Φεβρουαρίου, η διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε το αίτημα της αντιπροσωπείας να γίνει δικαιοποιητική συνεδρία στα πλαίσια τη Διατλαντικού Διαλόγου των ομοθέτων από 19 μέχρι 21 Ιουνίου στην Κροατία, τη χώρα της Προεδρίας, στο Ντουμπρόβνικ, βάσει της νέας σύνθεσης ε, της αντιπροσωπείας μετά το Brexit, η ποσόστοση των μελών που μπορούν να ταξιδέψουν θα, γίνουν, θα ε, υπολογιστούν εκ νέου τα ποσοστά και θα ενημερωθούν δεόντως τα μέλη. Έχουμε συνεδρίαση αντιπροσωπείας εις Washington και ο Στεφανούτα μόλις επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μας πει τις εντυπώσεις από τη συνεδρίαση του κόμματος στην Άιουα. Σημείο 4. Εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό, όπως ανέφερα, πρέπει να σεβαστούμε γεωγραφική ποικιλομορφία και την ισότητα των φύλων. Η πρώτη αντιπρόεδρος πρέπει να είναι γυναίκα και από χώρα εκτός Ρουμανίας πρέπει να είναι πλήρε μέλο, τακτικό μέλος αντιπροσωπεία και να έχει συμπληρώσει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων και τη δήλωση τη σχετική με τον κώδικα δεδειγμένης συμπεριφορά. Να ανακοινώσω τα ονόματα των αναπληρωτών που συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Έχουμε τον κατάλογο. Ετοιμάζεται ο κατάλογος. Ας έχουμε λοιπόν την υποψηφιότητα υποψηφιότητα για την εκλογή πρώτου αντιπροέδρου. Ορίστε. Προτείνω. Τη μία πέτρα κομπαρανάτσε. Επιφανές μέλος της Επιτροπής και αγαπητή συνάδελφο. Η υποψήφια δέχεται να είναι την υποψηφιότητα αυτή. Ναι. έχετε κάνει τα δέοντα για τα οικονομικά και το δοντολογικό κώδικα. Όπως βλέπετε από την ιστοσελίδα, ναι, έξοχα λέει ο πρόεδρος. Ε, άλλες υποψηφιότητες. Ευχαριστώ. Αν έχουμε μόνο μία υποψήφια, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Μπορούμε λοιπόν διαβοής να την εκλέξουμε. Συγχαρητήρια στην κυρία Μία, Μία Πέτρα Κουμπούλα Νάτρι. Παρακαλώ να έρθετε να καθίσετε δίπλα μου. Congratulations. And we proceed smoothly. Προχωράμε λοιπόν, λοιπόν σημείο 5, ανταλλαγή απόψεων για τα φορολογικά με τον Benjamin Angel, διευθυντή από τη Γενική Διεύθυνση Tax UD τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τηλεδιάσκεψη. Τον βλέπω ήδη στην οθόνη. Να του στις Βρυξέλλες. Καλώ ήρθατε στην συνεδρίαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Ο διευθυντή ο κ. Angel είναι για τον συντονισμό για άμεση φορολόγηση, οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια χαρά είναι η εικόνα και ο ήχος. Δεν χρειάζεται να πω σε κανένα από τους παρόντες πόσο σημαντικά είναι αυτά για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, τους επιχειρηματίες, για την φορολογική βάση, φορολογητέα βάση και την όλη η δημοσιονομική μας κατάσταση. 21 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες να εξασφαλίσει το ότι οι ψηφιακές επιχειρηματικές δραστηριότητε θα φορολογούνται δίκαια και φιλικά προς την ανάπτυξη. Πρωτοβουλία που στηρίζεται και από ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως θα θυμόσαστε. Αμερικα... Ο πρέσβης Σάντερλαντ, ο Αμερικανό προσκεκλημένο, είχε στεναρή θέση επί του θέματος και ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα, είναι ένα θέμα που αν προχωρήσει καλά, μπορεί να συμβάλλει σε οικονομική ανάπτυξη και σε καλές διατλαντικές σχέσεις. Αν δεν εφαρμοστεί καλά όμως, μπορεί να είναι αγκάθι στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Συμπεριλάβαμε διάφορα έγγραφα σαν ε, υπόβαθρο στους φακέλους σας. Πριν από τη συνεδρίαση πρέπει να είσαστε ενήμεροι φαντάζομαι και μπορούμε να αυξήσουμε τις πληροφορίες που περιέχονται εκεί συνομιλώντας με το διευθυντή τον κύριο Angel. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για την κουβέντα, για τη συζήτηση. Κύριε Angel, κάντε την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε να μιλήσω στην Επιτροπή σας. Αν με επιτρέπετε καταρχάς, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τον τρόπο λειτουργίας ε, της φορολογίας όπως συζητείται σε διεθνές επίπεδο και στη συνέχεια θα κάνω κάποια σχόλια για την κατεύθυνση που ε, ακολουθούμε και την πιθανότητα επίτευξη συμφωνία. Ο βασικός στόχο ε, τη συνεχίζόμενη συζήτηση είναι πολύ απλό. και δει να εξασφαλιστεί πω ε, η φορολογία θα γίνεται εκεί που παράγεται η αξία. Όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση με τους μεγάλους ομίλους και εταιρείε στην ψηφιακή κυρίω, ε, στο ψηφιακό κλάδο που έχουν μεγάλα κέρδη και τι περισσότερε φορέ δεν φορολογούνται στι χώρε που έχουν πολύ σημαντικό κύκλο εργασιών ή αν φορολογούνται πολύ λίγο. Ε, και στον ΟΥΣΑ, πάνω από 130 χώρες, υπάρχει αυτό το ε, πλαίσιο ε, που έχει δύο πυλώνες εκεί. Ο πρώτος πυλώνας είναι η αναδιανομή του κέρδους στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται πολυεθνικές εταιρείες, έτσι ώστε να υπάρχει δίκαιη κατανομή και επιμερισμός ε, του φορολογικού εισοδήματος που δημιουργείται ε, στη χώρα που δραστηριοποιείται η πολυεθνική. Το κατόφλι του κύκλου εργασιών που λαμβάνεται υπόψη είναι 750 εκατομμύρια, εκατομμύρια ε, ευρώ. Μόνο αυτές τις εταιρείες λοιπόν λαμβάνουμε υπόψη Εξετάζεται βέβαια το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα ονομαστικό σημείο αναφορά σε ένα national benchmark σε ό,τι αφορά την κατανομή. Πώ θα υπολογίσετε αυτό το σημείο τώρα αναφορά, Πολύ απλά. Θα βλέπει κανεί τι πωλήσει τη πολυεθνική και θα παίρνει ένα ονομαστικό 10% επιστροφή και θα αναδιανέμεται το 20% του κέρδους που υπερβαίνει το 10% αυτού του ονομαστικού συντελεστή. Και η αναδιανομή αυτή θα γίνεται μεταξύ όλων των χωρών που η πολυεθνική αυτή έχει αρκετή δραστηριότητα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συμπεφωνημένο τέτοιο όριο αναφοράς, benchmarks, ό,τι αφορά ε, το διακρατόμενο αυτό ποσό. Το σύστημα τώρα δεν θα περιοριστεί στο ψηφιακό κλάδο. Αυτό το οποίο είναι υποσυζήτηση είναι να αφορά εν γέννη τις πολυεθνικές, οι δύο τομείς που αποκλείονται, που εξαιρούνται από τις συζητήσεις, είναι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος με το επιχείρημα, το ξέρει και πολύ καλά η Επιτροπή ΕΚΟΝ, ότι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος ήδη ε, υποβάλλεται σε πολλές ε, ρυθμίσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα μέρη του κόσμου και το δεύτερο, δεν και τόσο σαφές ίσως, είναι η εξορρυκτική ε, βιομηχανία. Λόγω της τοποθέτησης κάποιων κρατών μελών του ωσά. Με ένα σκεπτικό που ομολογώ δεν το καταλαβαίνω απόλυτα δεύτερος πυλώνας. Είναι ένα φυσικό συμπλήρωμα του πυλώνα παρθμών 1. Και ο στόχος είναι να υπάρχει μια κατώτατη φορολόγηση του κέρδους, μια ελάχιστη φορολογία του κέρδους. Η συζήτηση, ως έχει αυτή τη στιγμή, φαίνεται να συγκλίνει γύρω σε ένα επίπεδο που αντιστοιχεί σε ένα που ισχύει ε, και σε κάποιο κράτος μέλος, 12,5%. Αυτό είναι το κατώτατο επίπεδο, 12,5%. Η αρχή είναι πολύ απλή. Αν η χώρα ε, που φιλοξενεί ε, μια πολυεθνική δεν ε, επιβάλλει επαρκή φορολογία, μπορεί η άλλη χώρα να επιβάλλει περισσότερο μέχρι ό,τι επιτευχθεί αυτό το ποσοστό και υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης του μέτρου αυτού με άλλη δέσμη μέτρων όπου δεν χορηγούνται φοροαπαλλαγές ή ε, μειώσεις, ώστε να ε, εξασφαλιστεί αυτό το κατώτατο επίπεδο. Οι έχουν ε, τη δική τους δέσμη μέτρων, guilty λέγεται, ενδιαφέρον, ενδιαφέρον είναι το ακρονίμιο αυτό. Και εκεί υπάρχει ένα κατώτατο επίπεδο αμερικανικής φορολογίας στο ξένο κέρδος ε, των πολυεθνικών ε, που έχουν την έδρα του στη ΣΥΠΑ. Στο κέρδος στην Αλοδαπή δηλαδή. Και υπάρχει και το σύστημα BIT. Τους αρέσει τους Αμερικανούς έτσι να διαλέγουν ε, εύγλωτα ακρονίμια. Για να μην υπάρχει διάβρωση βάσης σε περιβολικά μεγάλο βαθμό λόγω του συνδυασμού τέτοιων ελαφρύσεων και μειώσεων. Έτσι αντικαθρεπτίζονται και οι συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή πιστεύω και στο διεθνές επίπεδο. Πού βρισκόμαστε σήμερα. Στις αρχές της χρονιάς υπήρχε ελπίδα ότι θα έχει ε, βρεθεί ένα συμβεβασμό ε, στο λεγόμενο Inclusive Framework στο Παρίσι τον Απρίλιο, στο πλαίσιο του ΩΣΑ, δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό. Δεν υπήρξε συμβιβασμό, άρα γίνονται νέες προσπάθειες με στόχο να υπάρξει συμφωνία εν ώψη της νέας συνεδρίασης ε, του Ιουλίου στο Βερολίνο. Δεν είναι σαφές αυτή τη στιγμή κατά πόσον θα βρεθεί μια συμβιβαστική λύση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν αντιτεθεί ε, στεναρά στο πυλώνα 1 όπως συζητείτε και για αρκετό καιρό έχουν αφήσει έτσι να πλανάται η έννοια του face over που σημαίνει opting out μιας πολυεθνικής, δηλαδή δυνατότητα εξαίρεσης ε, ε, μιας ε, πολυεθνικής, που θα μπορεί να επιλέγει κατά πόσον θα δεχθεί να συμμετέχει ή όχι στο σύστημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί, διότι κάτι τέτοιο δυνητικά θα καταστρέψει το στόχο αυτού του συστήματος αν είναι κατά αλακάρτη η συμμετοχή στο σύστημα και θα ε, εξανεμιστεί το, το κέρδος που μπορεί να, να δούμε. Θα δούμε κατά πόσον θα μπορούσε να συμπεριληφθεί αυτή η υπόσχεση δέσμευση εξέτασης ε, μιας ε, ασφαλούς ε, επιλογής safe δεν έχουμε κάτι ξεκάθαρο ακόμα, ούτε υπέρ ούτε κατά και αυτό μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και τα δεδομένα για τον πυλώνα 1. Είπα, ε, στηρίζουν πιο πολύ τον πυλώνα 2. Και κυρίως διότι έχουν ε, εγχώρια μέτρα που είναι ένα βήμα αρκετά ισχυρό προς την υλοποίηση του πυλώνα αυτού. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυστυχώς είναι διαιρεμένα σχετικός. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που δεν στηρίζουν τον πυλώνα 1 και κάποια άλλα κράτη-μέλη που δεν στηρίζουν τον πυλώνα 2. Συνολικά, όλα τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρείται ότι αυτό είναι σημαντικό. Να σημειωθεί δηλαδή πρόοδος και είναι προτιμότερο να υπάρξει μια διεθνής συμφωνία παρά συλλογή εθνικών μέτρων που θα οδηγήσει ουσιαστικά σε ένα πλαίσιο που δεν θα είναι καθόλου ομοιογενές και δεν θα είναι και αποτελεσματικό εν τέλει. Είναι πολύπλοκο να τηρήσουν τις φορολογικές απαιτήσεις πολυεθνικές. Μια διεθνής συμφωνία όμως σημαίνει ότι υπάρχει ε, προτεραιότητα σε αυτήν, ε, υπερτερή αυτή η διεθνή συμφωνία. Από την άλλη, αν θυμάστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πρωτό, προτείνει μια προσωρινή γρήγορη λύση, τη φορολόγηση του ψηφιακού κλάδου. Οι συζητήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Συμβουλίου τελμάτωσαν. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη όμως που έχουν θεσπίσει εθνικά μέτρα, τα οποία εμπνέονται απευθείας από αυτή την πρόταση στην αρχή της Κομισιόν. Γαλλία, Αυστρία, Ιταλία, Τσεχία, Ουγγαρία. Και σήμερα έχουμε μέτρα και στην Ισπανία, τη Σλοβακία και το Βέλγιο. Το πιο γνωστό που έγινε πρωτοσέλιδο είναι το γαλλικό μέτρο, γιατί ξέρουμε ότι προκάλεσε την αγανάκτηση των Αμερικανών ομολόγων. Σε δύο προτάσεις θα σας πω. Φορολογούνται, το ο κυκλοστρασιών των επιχειρήσεων όταν αυτός υπερβαίνει 25 εκατομμύρια στη Γαλλία και συνολικά ε, ανέρχεται σε 750 εκατομμύρια. Υπήρξε μία έρευνα ε, εμπορική σε χώριο επίπεδο στη ΣΥΠΑ που κατέληξε στο ότι είναι ένα μέτρο που στρεβλώνει την αγορά και είναι δυσανάλογο. Και αποφασίστηκε να ληφθούν αντίπεινα. Αυτό είναι όμως εγχώρια απόφαση. Δεν έχει δοθεί πράσινο φως σε δένες επίπεδο από τον ΩΣΑ. Απλά το Κογκρέσο καλείται, καλεί μάλλον την κυβέρνηση να ε, αυξήσει τους φορολογικούς δασμούς για μερικά προϊόντα. Ο φόβος μας είναι πως θα κάνουν κίνηση, είπα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει την υποστήριξή της στις γαλλικές αρχές και έχει ξεκαθαρίσει και στις Αμερικανικές αρχές ότι αν κάνει αυτή την κίνηση η κυβέρνηση Τραμπ θα ληφθούν μέτρα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως απάντηση στην κίνηση, τον είπα. Όπως ε, έχουμε δει βέβαια, έκτοτε υπήρξαν επαφές μεταξύ των Προέδρων Τραμπ και Μακρόν, όπου και συμφωνήθηκε κάποιο είδους εκεχηρία, ανακοχή επί του παρόντος, οι ΙΠΑ δεν εφαρμόζουν κυρώσεις ε, και οι γαλλικές αρχές έχουν αναστείλει την ίσπραξη του φόρου. Μέχρι στιγμής οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη συζητήσει ένα παρόμοιο μέτρο με αυτό που ε, έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες που είπα, Ιταλία, Τσεχία, Αυστρία, γιατί ε, μπορεί να δημιουργηθούν και εκεί δύσκολες συζητήσεις. Σε αυτή τη φάση είναι δύσκολο να πει κανείς πόσο πιθανή είναι η επιτεύξη διεθνούς συμφωνίας εντός του τρέχοντος έτους. Σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος. Δεν ξέρουμε αν επαρκεί όμως αυτή η πρόοδος για να καταλήξουμε υπάρχουν αρκετές πιθανότητες και δυνατότητες. Εμείς θέλουμε ένα φιλόδοξο αποτέλεσμα με έναν πρώτο πυλώνα που θα εξασφαλίζει τον επιμερισμό των κερδών και θα καθιερώνει το κατώτατο συντελεστή φορολόγηση. Η πρόεδρο Φόντερ Λάιεν και ο επιτρόπο Τζεντιλόνι τα έχουν πει ε, κατηγορηματικά ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει διεθνή συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταθέσει νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την πολύ σημαντική προτεραιότητα για όλους τους πολίτες, δηλαδή μια δίκαιη αποτελεσματική φορολόγηση του ψηφιακού κλάδου. Θα ε, ολοκληρώσω εδώ την εισαγωγή μου και με τα χαρά θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Πριν ξεκινήσουμε το διάλογο, να θέσω δύο ερωτήσεις. Ε, καταρχάς, η Βρετανία εισήγαγε κάποια σχετική φορολόγηση. Είναι αποτελεσματική και ποια ήταν η ανταπόκριση των Αμερικανών στη Βρετανική ε, κίνηση. Δύο, σε ποιους τομείς του θέματος λαμβάνεται απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πλειοψηφία και σε ποια σημεία χρειαζόμαστε ομοφωνία, για ποιες αποφάσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το πρώην κράτος μέλος μας συζητά την θέσπιση του νόμου αυτού, της φορολόγησης αυτής, αλλά δεν ισχύει ακόμα αυτός ο φόρος. Δεν υπάρχει ανοιχτά συζήτηση με τη είπα για αντίπεινα ε, έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα τι χρειάζεται όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων. Πρέπει να υπάρχει διεθνή συμφωνία στον ΟΣΑ. Νομικά αυτή η συμφωνία για μας δεν μπορεί να είναι κάτι απομονωμένο. Πρέπει να προταθεί η νομοθεσία για την ενσωμάτωση αυτής της συμφωνίας στο εθνικό δίκαιο. Η νομοθεσία σε αυτό το τομέα απαιτεί ομοφωνία, αλλά έχουμε την πεποίθηση ότι σε περίπτωση πολυμερών συμφωνιών, πολυεθνικών συμφωνιών, τα κράτη-μέλη θα έχουν συμβάλει στη σύναψη αυτής της διεθνούς συμφωνίας και εκεί μπορεί να επιτευχθεί ομοφωνία όσον αφορά τα μέτρα που ενσωματώνουν τη διεθνή συμφωνία αυτή ε, στον ΩΣΑ. Ο κύριος Τάγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι ερωτήσεις σας ήταν ακριβώς, ε, ήταν πολύ ευστόχες. Και έτσι απαντήθηκαν και κάποιες από τις δικές μου. Προ, προς τον Διευθυντή Αντζέλ ε, απευθύνω την ερώτηση, τον κύριο Ανζέλ. Λοιπόν, είμαστε κατά των φορολογικών παραδείσων. Αυτό είναι ο δεύτερο πυλώνα και συμφωνούν οι Αμερικανοί. Ο πρώτο πυλώνα είναι κατά των μεγάλων επιχειρήσεων. Και οι Αμερικανοί δεν συμφωνούν. Κατά την άποψή μου, τι μπορούμε να αναμένουμε. Συμφωνία στον ΟΣΑ για τον πυλώνα 2 και αν υπάρξει ίσως τύχη αποδοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλη την ομοφωνία, την αρχή της ομόφωνης απόφασης. Όμως, ίσως πρέπει να είμαστε υγιώς σκεπτικιστές όσον αφορά τη συμφωνία στον πυλώνα 1. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα των συζητήσεων σε βάση του ΟΣΑ που θα οδηγούσαν σε απόπειρα πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω να ακολουθήσουμε το, δρόμο, το δικό μας δρόμο, ούτως υπήν, τη δική μας πορεία. Κύριε Τάγκ, η ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Είμαστε κάπω πιο αισιόδοξοι όσον αφορά τι διαπραγματεύσει όσα ήμασταν πριν από ένα χρόνο, μισό χρόνο, μετά τη διαφωνία Γαλλία-ΗΠΑ. Ήμασταν πιο αισιόδοξοι παλιά. Τώρα όμω έχουν περάσει σε δύσκολη φάση οι συζητήσει, αλλά τρέφουμε ελπίδε. Δύο ερωτήσει. Η πρώτη σχετίζεται με τις έξω του Μάρεκ Μπέλκα. Έχουμε διαπραγματεύσεις, διότι έκανε για τον DST προτάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και δώσαμε το μήνυμα ότι είμαστε σοβαροί, ότι θέλουμε να φορολογήσουμε τις μεγαλύτερες ε, εταιρείες. Και τελικά οθήσαμε τους Αμερικανούς να έρθουν ε, στο τραπέζι. Και αυτοί είπαν ότι και ασκούμε πιέσει πάνω τους. Μήπως πρέπει να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα για να θεσπιστεί το DST ή να πιέσουμε για τις διαπραγματεύσεις. Για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Να προτείνουμε κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προτείνουμε ότι το Δεκέμβριο 2020 θα κάνουμε μια πρόταση όσον αφορά το φόρο ψηφιακών υπηρεσιών. Την πρόταση του ΩΣΑ τη βλέπω με πολύ θετικό μάτι, διότι ο πυλώνας 1 θεσπίζει στοχευμένες αρχές, προορισμό, την αρχή του προορισμού. Και ήταν η αρχή που χρησιμοποίησαμε στο σύστημα CCTV Καλή κατεύθυνση. Τα αποτελέσματα, τα πρακτικά, ποια θα είναι. Θα ωφεληθεί όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα, φαντάζομαι, Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε αξιολόγηση αντικτύπου, δεν είδα τους αριθμούς. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία. Κύριε Έιντζελ, για τους φορολογικούς παραδείσους συμφωνώ, είναι πολύ σημαντικό μέχρι 53 ευρώ στον κόσμο βρίσκονται σε φορολογικούς παραδείσους. Σκεφτείτε τι μπορούμε να κάνουμε 53 εκατομμύρια ευρώ. 3 εκατομμύρια. Κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξεκινώ με την ερώτηση του Πρωθυπουργού του κυρίου Μπελκά. Το δυσκολότερο ερώτημα θέσατε. Δηλαδή, τι αποτελεί επιτυχία και τι αποτυχία στις διαπραγματεύσεις του ωσα Συμφωνώ. Το υπονοούμενο πίσω από την ερώτησή σας είναι ότι ελοχεύει κάποιος κίνδυνος. Δηλαδή να καταλήξουμε σε κάτι που έχει την ετικέτα διεθνούς συμφωνίας, αλλά δεν θα είναι τόσο ισχυρή όσο θα θέλαμε. Θα είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Δεν μπορώ να απαντήσω σήμερα την ερώτησή σας. Είναι πολιτική αξιολόγηση που αφορά τον πίτρο Τζεντιλόνη και την Πρόεδρο Βοντελάιν. Πρέπει να πάρουν απόφαση βάση της ε, συμφωνίας που θα επιτευχθεί. Να αποφασίσουν κατά πόσο αρκεί η συμφωνία, αν μας ωφελεί αν θεωρούμε ότι έχουν καλυφθεί οι ανησυχίες μας. Σήμερα, αν αυτό που έχουμε μπροστά μας, αν μας ικανοποιεί, ε, ότι δεν εγκρίνεται ο πυλώνας ένα, αν αυτά που συζητούνται στον ΩΣΑ συνεχιστούν να συζίζονται, προτεραιότητά μας θα είναι να εφαρμοστούν αυτά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σωματωθούν και στα εθνικά δίκαια. Τώρα, αν αυτό θα γίνει ή δεν θα γίνει, δεν το ξέρω. Υπάρχουν κάποιοι στον όσα, κάποια κράτη-μέλη, κάποια κράτη στον Νόσα που λέτε ότι οι λεπτομέρειες των υπολογισμό του κέρδους και να γίνει αναδιανομή είναι θέματα προς επανεξέταση και αν να πάρουμε το 20% του κέρδους να παίρνουμε ένα ονομαστικό, να θεωρήσουμε ένα απόδοση 10% ή να πάμε πάνω από 20%. Αυτό προσπαθούμε να αποφασίσουμε. Ίσως τέτοιες δυσκολίες αντιμετωπίσουμε. Γιατί μπορεί να καταλήξουμε ότι αυτή η περιπτώση συμφωνία στον πυλώνα 1 που πρακτικά δεν θα έχει πολλά αποτελέσματα. Στην πράξη, ο όγκος των κερδών που θα ανακατενεμηθεί σε όλο τον κόσμο πιθανότατα θα είναι διψήφιο σε αριθμός για τον πλανήτη. Διψήφιος αριθμός ε, για όλο τον πλανήτη μάλλον δεν είναι εντυπωσιακό νούμερο, χρειάζεται πολιτική απόφαση. Όταν θα υπάρχει καθαρό αποτέλεσμα και διεθνής απόφαση στο κατά πόσο ικανοποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση με το αποτέλεσμα. Ή αν θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι χρειάζεται να τεθεί πιο φιλόδοξος στόχος. Δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε όμως. Αν υπάρξει διεθνές αποτέλεσμα, θα σκηθούν ισχυρότατες πιέσεις να συμμορφωθούμε. Από παντού, από όλους τους εταίρους θα μας πιέσουν. οποιαδήποτε μέτρα που ξεπερνούν πέρα, πέρα, πέρα από αυτό το όριο θα θεωρούνται ότι υπονομεύουν τη Διεθνή Συμφωνία. Γι' αυτό λέω ότι η πολιτική συζήτηση θα πετηθεί. Γιατί αυτή η απόφαση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η ερώτηση του κύριου Τάγκ. αν πρέπει να αναζωογονήσουμε το φόρο των ψηφιακών υπηρεσιών και να θέσουμε σταθερή, συγκεκριμένη μάλλον προθεσμία. Αναζωογόνηση του, του φόρου ψηφιακών υπηρεσιών είναι περισσότερο στα χέρια των 100 μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πρόταση, είναι επιτάπητος, είναι στο Συμβούλιο η πρότασή μας. Ο Επίτροπος Ζεντιλόνη και η πρόεδρος Βοντελάιν είπαν ότι αν μέχρι το τέλος του χρόνου δεν έχουμε πρόοδο στον ΩΣΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις, θα εξετάσει τον δεχόμενο υποβολής προτάσεων. Αυτό είναι το ίδιο με το θέμα που συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό Μπαλκά στο τέλος θα μπορέσουμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα κατά πόσο υπάρχει συμφωνία ή όχι και αν ναι, αν είναι ικανοποιητική συμφωνία. Δεν το γνωρίζουμε, άγνωστο. Αυτή είναι η ειλικρινή απάντηση ότι δεν γνωρίζω. Ποια είναι τα πραγματικά αποτελέσματα. Διανύμαμε κάποια στοιχεία εδώ και κάποιους μήνες στα κράτη-μέλη. Ήταν αρχική υπολογισμή αυτή. Βάση των, των στοιχείων που συζητούσαμε τότε. Οι διεθνείς συζητήσεις μεταβάλλονται συνεχώς, οπότε επανειλημμένα ξεκινάμε από το μηδέν, ε, προσαρμόζουμε τους υπολογισμούς, είμαστε σε επαφή με τον ΩΣΑ. Ανταλλάσσουμε στοιχεία. Συζητάμε προσεγγίσεις όσον αφορά τον καλύτερο υπολογισμό των αποτελεσμάτων του πυλώνα 1 και του πυλώνα 2. Θα δημοσιεύσουμε αποτελέσματα, πιθανότατα, της συνεχιζόμενης προσπάθειας κάποτε πριν το καλοκαίρι. Δεν έχω ακόμα κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, διότι οι εργασίες συνεχίζονται. αν μιλήσει κανείς γενικά όσον αφορά τον αντίχτυπο για τα κράτη-μέλη, αναπόφευκτα θα έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Δεν θα επικρατεί ομοιομορφία συναρτήση του πυλώνα. Ο πυλώνας ένας, ένα ως έχει θα οδηγήσει σε μείωση των φορολογικών εσόδων των κρατών μελών που έχουν μεγάλους ε, οικονομικούς κόμβους ο πυλώνας 2 θα αυξήσει όμως το φορολογικό έσοδο των κρατών μελών με τα μεγάλα οικονομικά κέντρα. Τώρα για τα περισσοτερα κάτι κράτη-μέλη θα γίνει. Θα πρέπει να έχουμε τους δύο πυλώνες. Θα ήταν θετικό με τους δύο πυλώνες στην όλη εικόνα δεν θέλω να ρίξω κάποιο νούμερο σήμερα. Θα ήταν αμφισβητήσιμα αυτά τα στοιχεία τα αριθμητικά, εφόσον όπως σας είπα συνεχίζονται οι εργασίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος να έχει μια ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω και ένα σχόλιο, καταρχάς, πριν την ερώτηση. Το σχόλιο είναι ότι οι πιθανότητες να υπάρξει συμφωνία έχοντας υπόψη τις εκλογές της ΕΕ, και το πώς χρηματοδοτεί την πολιτική εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξε. Για τον πρώτο πυλώνα, ε, το ερώτημά μου που είναι λίγο τεχνικό. Για να υπολογιστεί η προστέμενη εξά το κέρδος δηλαδή και να περάσουμε το 10% ή το 20% αυτό το κατόφλι Χρειάζονται και τα έσοδα αλλά και ε, το κόστος. Πρέπει να υπολογιστούν και οι δύο παράμετροι σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Είναι έτσι καλά, το έχω καταλάβει και αν ναι, ποιες είναι οι αρχές λογιστικής κόστους που εφαρμόζονται διεθνώς. Υπάρχει αναρμόνιση, υπάρχει εποπτεία ρύθμιση. Αν μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ για το πρώτο. Οι εκλογές σίγουρα δεν διευκολύνουν μια γρήγορη συμφωνία και η σημερινή κυβέρνηση, τον είπα όπως γνωρίζετε, ε, κάποιες φορές ε, φάσκει και αντιφάσκει. Οπότε θα είναι δύσκολο να υπάρχει συμφωνία σε επίπεδο ΩΣΑ. Θα εξαρτηθούν πολλά από τι εκλογέ του Νοεμβρίου. Σε αυτή τη φάση καμία πρόβληψη δεν μπορεί να γίνει για την τελική στάση της ε, Αμερικανικής κυβέρνησης. Ε, θα ήταν απλή κασία. Όπως είπε όμως και ο κύριος Τάγκ, συμμετέχουν ενεργά στηρίζουν ενεργά τον πυλώνα 2. Εμείς απλά πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να τους κάνουμε να υποστηρίξουν και τον πυλώνα 1. Γιατί έχουμε τη θέση μας για τον ασφαλή λιμένα που θα υπονομευθεί. Και σίγουρα οι επαφές με το Κογκρέσο ε, θα ήταν κάτι θετικό αν μπορείτε και εσείς να περάσετε το μήνυμα και να μας υποστηρίξετε. Ότι χρειαζόμαστε δηλαδή έναν αξιόπιστο πυλώνα 1. Τώρα, ως προς τις ε, συνέπειες, τους κανόνες λογιστικής. Αν υπάρξει την συμφωνία, θα υπάρξει ε, και μία πληθώρα θεμάτων στα οποία θα πρέπει να δώσουμε μία συνέχεια. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα έχουμε λύσει τα θέματα με τα λογιστικά πρότυπα, αλλά αν μιλάμε για παράδειγμα για ελάχιστη φορολογία, είχαμε κατά το παρελθόν κάνει κάποια συζήτηση, χωρίς δυστυχώς όμως ακόμη να έχουμε καταλήξει κάπου. Και φυσικό επακόλουθο είναι να ξαναρχίσει αυτή η συζήτηση. Φορολογική βάση είναι ένα θέμα που θα ανοίξει. Αν έχουμε αυτό το κατώτατο στελιστό 12,5%, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ένα κοινό όριο αναφορά, ένα benchmark. Ποια είναι η φορολογική βάση στην οποία εφαρμόζουμε αυτό το 12,5%. Αν υπάρξει διεθνή συμφωνία, θα είναι αυτή μια σημαντική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να σημειώσει πρόοδο πάνω σε ε, φακέλους που εκκρεμούν εδώ και καιρό. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να ανανεώσουμε και τις προσπάθειές μας για να καταλήξουμε σε μια κοινή προσέγγιση σίγουρα θα υπάρξουν επιπτώσεις σε διάφορους κλάδους. Θα ήταν πρόωρο όμω ε, να προβώ σε λεπτομερή ανάλυση από τη στιγμή που δεν ξέρουμε ακόμα ε, τι θα αποφασίσει η Αμερικανική κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις, λέει ο Πρόεδρος, αν όχι, να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος ε, όλη τη αντιπροσωπεία, κύριε Έντζελ, για το χρόνο που μα διαθέσατε, για τι απαντήσει σα και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν οι συναδελφοί μου με το ότι οι πολίτες πραγματικά απαιτούν ένα σύγχρονο σύστημα προσαρμοσμένο στη σημερινή πραγματικότητα, συμβατό με τη μορφή που έχει η παγκόσμια οικονομία και ένα σύστημα που πρέπει να είναι δίκαιο και αποτελεσματικό. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να προσθέσω ότι κατ' εμέ αυτό είναι και ένα από τα βασικά, από τα μείζωνα ζητήματα της εποχής μας, που μπορεί να φαίνεται τεχνικό, όμως στην ουσία έχει να κάνει και με τη ρίζα της ανομίας στην κοινωνία, δηλαδή την αντίληψη ότι τον πλούτο τον έχουν στα χέρια τους ιδιώτες και οι μεγάλοι όμιλοι, οι μεγάλες εταιρείε δεν ε, συνεισφέρουν αναλογικά στις υποδομές, ε, τις ε, φυσικές και ανθρώπινες που χρησιμοποιούν. Ούτε ανταγωνίζονται δίκαια αλλήλους. Αν κάποιος δραστηριοποιείται σε επίπεδο ε, πληρώνει ε, αλλά όχι μεγάλες πολυεθνικές που έχουν ε, δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο και πληρώνουν ελάχιστα. Θα πρέπει λοιπόν να αποκαταστήσουμε την αίσθηση του δικαίου στις παγκόσμιες συναλλαγές γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς θα το κάνουν οι δημαγωγοί, οι λαϊκιστές και με λάθος τρόπο και προκαλώντας μεγάλες ζημιές. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα κυρία Διευθυντά. Εκτός μικροφώνου, πρόεδρος. Εκτός μικροφώνου, πρόεδρος, δεν ακούγεται. Uh, for uh, translations into Greek. Είχε ζητηθεί μετάφραση ελληνικά, πολωνικά, γαλλικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπω όμως ότι αυτοί που τη ζήτησαν δεν παρίστανται. Αυτό να το λάβουν υπόψη μας παρακαλώ. Οι πολίτες ζητούν από εμάς να χρησιμοποιούμε φιδωλά τα χρήματα των φορολογουμένων. Άρα να δαπανούμε χρήματα σε αχρία στη διερμηνία ε, είναι περί τη δαπάνη. Έρχομαι στο έξι που είναι τα διάφορα. Ο κύριο Στεφάνουτα μόλις γύρισε από την Άιωβα. Για παρακαλώ να μας πείτε τι που αποκομίσατε. Ναι, φαντάζομαι όλοι καίγεστε να μάθετε τι έγινε στην Άιωβα. Θα ήθελα να σας πω λίγο πράγματα για το πλαίσιο που μπορεί να είναι και χρήσιμο για όλους. Ε. Ήμουν στην αντιπροσωπεία του κόμματος και πρέπει να σας πω ότι πέραν της επίσημης αντιπροσωπείας υπάρχουν και κάποιες ε, αντιπροσωπείς κομμάτων ή ομάδων ε, που επισκέπτονται τους πολιτικούς του συμμάχους ε, στις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, πηγαίνουν κάποιοι σε συνέδρια των δημοκρατικών, των ε, συντηρητικών που διαλέγουν να δίνουν το χρήσμα και έχουμε τον Ιούλιο τους δημοκρατικούς και οι Ρεπουμπλικανοί νομίζω είναι τον Αύγουστο. Παρακαλώ συζητήστε μήπως κάποιος από κόμμα σας θέλει να μεταβεί με μια αντιπροσωπεία. Είδαμε λοιπόν με το Αιώβα Κόκκους, παρατηρήσαμε την εκλογική ε, διαδικασία, μια παλιά διαδικασία. Αυτό το κόκκους τι θα πει, είναι κάποιοι οποίοι έρχονται ε, και πηγαίνουν και στείνονται σε μια γωνία της αίθουσας. Είναι ενδιαφέρον το βλέπει κανείς, αλλά τελικά όλο αυτό κατέληξε σε χάος, γιατί το σύγχρονο στοιχείο δεν λειτουργήσε οι εφαρμογέ, στο application και η δημοκρατική, σε ό,τι αφορά τη δημόσια εικόνα, είχαν πλήγμα. Του στήχησε. Και ακόμη και ο πρόεδρο στην ομιλία του για την κατάσταση τη Ένωση την ίδια ημέρα. Το ε, εκμεταλλεύτηκε το ότι δεν μεταφέρθηκαν σωστά τα αποτέλεσματα από του δημοκρατικού δηλαδή. Να έρθω σε δύο-τρία σύντομα στοιχεία. Μεγάλη προσέλευση πολύ ενδιαφέρουν γιατί αναγνωρίζουν ότι είναι, για, ότι είναι σημαδιακή η χρονιά, είναι απτό αυτό. Ο Τραμπ μιλάει για το πλήθος που τον συνοδεύει και που είναι υψηλό, ναι, αλλά και στους δημοκρατικούς είχαμε πολλούς. Το κόστος όμως για τους δημοκρατικούς δεν ήταν καλό. Ο Σάντες και ο Μπούντιτσιτς είναι, ε, δίνουν μάχη στήθος με στήθος. Το θέμα είναι ποιος δίνει τα πιο πολλά χρήματα. Αρχίζουν τώρα να επενδύουν στον Μπούτιτζιτς. Ο Σάντερ είναι ο πιο πιθανός υποψήφιος για τους δημοκρατικούς με βάση τις δημοσκοπήσεις και δύο κόκκους έχουν επιβεβαιώσει ε, αυτή τη θέση. Άρα, χωρίς να θέλω κι εγώ να προβασικασίες, ε, η τάση τουλάχιστον είναι αυτή, θα δούμε πώς θα πάει η κούρσα τον, ε, το, το φθινόπωρο, θα είναι ενδιαφέρον. Τώρα, μεταξύ των Ρεπουμπλικανών έχει τη μεγαλύτερη δημοτικότητα ο Τραμπ, 49% φωτοεξελέγει. εξελέγει. Πολύ ψηλά ποσοστά θα έλεγα. Και ως Ευρωπαίος βουλευτής και μέλος της αντιπροσωπείας, δεν άκουσε ούτε μια φορά τη λέξη Ευρώπη. Ούτε και πολλά θέματα δεν ενδιαφέροντα. Τα δύο μόνο που αναφέρθηκαν ήταν από τον υποψήφιο Μπούτιτζιτς που είπε ότι αν γίνει πρόεδρος θα περιορίσει τις θητείες για σε τρία έτη. Αυτό κατ' εντολή του Κογκρέσου, αλλά περιορισμένη διάρκεια. Και ο Σάντερς είπε για την κλιματική αλλαγή ότι θα μιλήσει με Κίνα και Ινδία για να συμφωνήσουν. Μέχρι στιγμής αυτά όλοι μιλούν για υγεία, παιδεία, εσωτερικά θέματα και κλιματική αλλαγή. Περιέργως, όχι και με τόσο διεθνή πρόπτικη για το εμπόριο, Κανείς δεν μίλησε για το εμπόριο από μακριά. Κάποιες φήμες υπάρχουν ίσως. Ένα καρουσέλ δεν το ξέρουμε. Θα δούμε. Πάντως ήταν μεγάλη εμπειρία να δω τους υποψηφίους, από τι στόφα είναι φτιαγμένοι και έτσι να ακούσω και τις απόψεις τους. Ευχαριστώ. Any other business? Στα διάφορα. Α, δεν έχουμε. Να σας πω για τους δασμούς ότι η αντιπροσωπεία ίντα στην οποία συμμετέχω θα πάει στη Ουάσιγκτον σε δύο εβδομάδες και Μπέτ Λάγκε προεδρεύει. Θα έχουμε πολλές επαφές για τα θέματα των δασμών σε 15 μέρες. Ευχαριστώ. Θα ξανασυνεδριάσουμε την ίδια μέρα στο ίδιο μέρος στις 12 Μαρτίου. Πέρασε συνεδρίασης.